Καθίστε παρακαλώ αγαπητοί συνάδελφοι. Θα γίνει τώρα η υπογραφή της διαθεσμικής συμφωνίας μεταξύ του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Κομισιόν για την καλύτερη νομοθεσία και θα ήθελα εδώ να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για τα προς τα άλλα θεσμικά όργανα τη Ευρώπη της Ευρώπης την κυρία Ίνες Πλασά, Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το γεγονός ότι είστε εδώ παρούσα και έτοιμοι να υπογράψετε αυτήν την συμφωνία. Και θέλω να ευχαριστήσω και τη Λουξεμβουργική Προεδρία και τον κύριο Νίκολα Σμιτ για την δική του προσπάθεια για να μπορέσει να γίνει δυνατή αυτή η υπογραφή και συγχρόνως θέλω να ευχαριστήσω τον Επίτροπο τον πρόεδρο της Επιτροπής κύριο Γιούγκερ που με τι προσπάθειε τη Κομισιόν και ιδίω και του κ. Φραντ Τίμερμαν, του αντιπρόεδρου τη Κομισιόν, επένδυσε πάρα πολύ χρόνο σε αυτέ τι διαπραγματεύσει. Και θέλω να ευχαριστήσω και έναν συνάδελφο βουλευτή, ο οποίο έπαιξε σημαντικό ρόλο για να μπορέσει να γίνει πραγματικότητα αυτή η συμφωνία. Και πιστεύω ότι με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε ένα σημαντικό ορόσημο στις θεσμικέ μας σχέσεις με την Κομισιόν και την ε, το Συμβούλιο θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Γκίφιε Φερχόφστατ για το έργο του προς την κατεύθυνση αυτή και παρακαλώ τώρα να έρθουν οι εκπρόσωποι για να λάβουν μέρος στην τελετή υπογραφής. Πρώτα η κυρία Χένις Πλάσερτ.